Κυρίε και κύριοι, είναι 5 και 7. Έχουμε ψηφοφορίες, γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα γεμάτη με ακροάσεις των υποψηφίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η συνεδρίαση με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος το λόγο. Περνάμε λοιπόν αμέσως στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Στη γραπτή διαδικασία της 19 Σεπτεμβρίου, οι συντονιστές αποφάσισαν καταρχάς την έγκριση μιας έκθεσης πρωτοβουλίας για την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των Φίλων και την έγκριση μιας αποστολής στην Κροατία από τις 9 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019. Στην αποστολή θα μεταβούν 7 μέλη, δηλαδή κάθε πολιτική ομάδα θα εκπροσωπηθεί. Μετά από τις ανακοινώσεις περνάω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στις ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό το 2020 όλα τα τμήματα. Η ηλεκτρονική θα είναι η ψηφοφορία, γι' αυτό λοιπόν θα σας ρωτήσω αν έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία και θα ρωτήσω την εισηγήτρια κυρία Φιτζέραλτ αν θα ήθελε να πει δύο λόγια πρωτού ψηφίσουμε. Όχι. Θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Ωραία. Νομίζω... Νομίζω ότι όλα έχουν συζητηθεί στις διάφορες συνεδριάσεις. Είναι σαφές το τι επιλογές έχουμε, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να τοποθετηθείτε αλλά προχωράμε αμέσως στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία, αν δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας, προσπαθήστε σε ένα άλλο. Αν δεν λειτουργεί ούτε εκείνο, τότε μάλλον θα έχει πρόβλημα η κάρτα σας. Ίσως την έχετε τοποθετήσει λάθος. Όχι. Ωραία λοιπόν, θα σας έχω υπόψη σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο επόμενο πρόβλημα και θα μετρήσω την ψήφο σας για το ΕΛΚ. Ωραία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 1 με 19 ψήφους υπέρ. Ψηφίζεται υπέρ. Εντάξει, τότε να το δείξετε με ανάταση του χεριού και θα μετρήσω. Ωραία, πέρας λοιπόν. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία με 19 υπέρ και 6 κατά. Περνάμε στην επόμενη. Τροπολογία 18. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ψηφοί υπέρ, 4 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, μάλλον λειτουργεί το μηχάνημά σας. Εγκρίνεται λοιπόν με 19 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 της κυρίας Βάνα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 ψηφί υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Τροπολογία 27. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 0 κατά. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Τροπολογία 48. Α, όχι, με συγχωρείτε. Καταπίπτει αυτή η τροπολογία. Περνάμε στην 32 της κυρίας Νόχλη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 20 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 33 της κυρίας Βάνα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 22 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, 39. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 22 ψήφους υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ και 3 κατά. Τροπολογία 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 46 της κυρίας Βυσνιεύσκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 22 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56 της κυρίας Fitzgerald. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58, κύριο Τζόνς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με 17 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Τροπολογία 60. Τζάκι Τζόνς, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19 ψήφιτα υπέρ, 5 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της κυρίας Νόχλη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ 3 κατά εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά β' α, τοπολογία 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7 της κυρίας Βυσνιεύσκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Μας λείπει ένας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Και τροπολογία 12, κύριε Βυσνιεύσκα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελειώσαμε. Πρόκειται για προϋπολογισμό. Θα περάσουμε λοιπόν στο τέλος της ε, σημερινής ψηφοφορίας. Είδατε πως ήμασταν πολύ γρήγοροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την συγκίτρια. Τη συγχαίρω για την επικοδομητική συνεργασία που είχε με όλους τους σκιώδεις. Α, ναι, και έχω κάτι προς ενημέρωση. Μη φύγετε, μη φύγετε, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έκανα ένα λάθος. Ο προπολογισμό γίνεται πάντα χωρί τελική ψηφοφορία, όμω εδώ πρόκειται για γνωμοδότηση και η γνωμοδότηση πρέπει να ολοκληρωθεί με τελική ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν μη, μη μου φύγετε, παραμείνετε εδώ. Βιάστηκα. Γιατί είχα συνηθίσει από τον προπολογισμό που απλά ψηφίζαμε. Όμως στις γνωμοδοτήσεις έχουμε τελική ψηφοφορία η οποία άρχεται. Σα δίνω χρόνο να ξαναχρησιμοποιήσετε τις κάρτες και με συγχωρείτε. Ενεργοποιηθήκατε, μάλιστα. Μας λείπει κάποιος. Έχετε βάλει όλε τι κάρτες. Ωραία. Πέρα ψηφοφορία, όλοι ψήφισαν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, 19 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τα διάφορα. Εάν δεν υπάρχει κάτι προς συζήτηση, έτσι νομίζω, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 6 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Και θα περάσουμε τώρα στις συνεδρίες των συντονιστών. Ja, alles gut. ich war